Yes, we have to start the meeting. We are already... Ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε ήδη αργήσει λίγο. Δεν ξέρω, δεν έχουν ξυπνήσει οι ευρωβουλευτές φαίνεται. Μια που κάποιοι από εμά όμως έχουμε ξυπνήσει, ας αρχίσουμε. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω εδώ τον ε, κύριο Τόμ Μπέβερς που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης ΕΜΚΟ και τον κύριο Τόμας Ντομινίκ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, CPC. Θα δώσω πρώτα το λόγο λοιπόν στον κύριο Μπέβερς και νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ στην Επιτροπή αυτή είμαστε εξοικειωμένοι με την οργάνωσή σας, την θέση σας στο σύστημα, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα για τους νέους ευρωβουλευτές, αν μη τι άλλο, να μας εξηγήσετε λιγάκι ποιες είναι οι σχέσεις μας και ποια είναι η δικιά σας θέση στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Από τότε που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 148 της Συνθήκης Επιτροπή μας το 1998, η ΕΜΚΟ είναι το κύριο προπαρασκευαστικό όργανο που προετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Απασχόλησης, το ΕΦΣΚΟ. Ετοιμάζει τη στρατηγική, στρατηγική και της Λισαβόνας που τώρα έχει γίνει του 2020 και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε 17 χρόνια εμπειρίας λοιπόν στο συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών και όσον αφορά τη σύγκληση και όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών, δεδομένου βέβαια ότι δεν μπορεί ένα μοντέλο να ταιριάζει σε όλους. Υπάρχουν βέβαια και στο εξάμεινο κάποια στοιχεία κλειδί. Αυτή τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποία έχει ετοιμάσει την δικιά της έρευνα και τις εκθέσεις της για τις χώρες μέλη. Ετοιμάζονται τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και κάποια μηνύματα. Έτσι και το ΕΠΣΚΟ θα έχει την δικιά του συνεισφορά στο Εαρινό Συμβούλιο. Έχουν υποβάλει και χώρες μέλη τα προγράμματα αναθεώρησής τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα εκδώσει τις δικές της συστάσεις, θα τις συζητήσουμε, δεχομένως θα τις τροποποιήσουμε πριν αποτελέσουν συστάσεις για το Συμβούλιο τον Ιούνιο τον Ιούλιο. Επίσης όλο το χρόνο παρακολουθούμε τι έχει γίνει με τις συστάσεις έτσι ώστε να έχουμε μια πολύπλευρη άποψη για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί είναι μια δουλειά που κάνουμε με ιδιαίτερη προσοχή και, έχουν, και έχουμε επενδύσει πολύ σε αυτή. Η προσέγγιση μας διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη των πολιτικών συζητούνται σε βάθος, με ανοιχτό πνεύμα και βάσει στοιχείων καταλήγουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Φέτος, το εξάμεινο, εξετάζουμε και το Δεκέμβριο μάλλον το κάναμε, ε, το τι γίνεται με την ανεργία των νέων να παρακολουθήσουμε πώς εφαρμόζεται η εγγύηση για τους νέους. Θα ακολουθήσουν και νέες αναθεωρήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα συνεργαστούμε και με άλλες επιτροπές, όπως εκείνη της εκπαίδευσης για τη διαβίου κατάρτιση και με την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, μεταξύ άλλων για τη φορολογία. Βάσει των αθωρήσεων αυτών, το 2014 τροποποίησαμε διάφορες από τις συστάσεις που έστειλε η Επιτροπή σε μας και όλες αυτές οι αλλαγές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο. Επίσης, είχαμε ενισχυμένη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα σημεία κλειδί. Διαβουλευτήκαμε μαζί τους. Από την αρχή της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Επιτροπή μας είναι πεπισμένη ότι η δουλειά μας πρέπει να είναι καλύτερη ποιότητα όσον αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις μας πρέπει να βασίζονται σε συμπεράσματα και σε πρόθεση πολιτικών. Έχουμε επενδύσει πολύ όπως σας είπα και η επένδυση μας αυτή έχει αποδώσει. η αποφάση του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πλέον είναι πιο ισχυρές. Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία η οποία βέβαια απαιτεί προσαρμόσεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου μετά από τις συστάσεις της δικιάς μας Επιτροπής και της Κοινωνικής Επιτροπής με την οποία θα συζητήσετε αργότερα. Όπως θα γνωρίζετε επίσης είμαστε στα τελευταία στάδια της διάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής για το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αλλαγές στη μηχανική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προσβλέπουμε σε ένα τελικό πακέτο προτάσεων με σχέδιο για νέες κατευθυντήριες γραμμές και για την οικονομική πολιτική. Είχαμε την ευκαιρία να προσφέρουμε στο Συμβούλιο ΕΦΣΚΟ την κοινή γνωμοδότησή μας από τις δύο επιτροπές μας που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο από το Συμβούλιο και, εξετάζουμε, και θα εξετάσουμε το πακέτο όταν θα τα έχουμε συνολικά. Θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτές και κυρίως της απασχόλησης αποτελούν πολύ βασικό στοιχείο της αναθεώρησης γιατί καθορίζουν έναν ευρύ προσανατολισμό για την ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης. Είναι καθήκον της δικιάς μας Επιτροπής και θα αρχίσουμε τις συζητήσεις όταν θα έχουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ακούσουμε και τις απόψεις της δικιάς σας Επιτροπής βεβαίως και ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς στην ΕΜΚΟ έχουμε διασαφηνίσει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς. Πρέπει να επιβεβαιωθεί ο στρατηγικός ρόλος που έχουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει επίση να είναι πλήρε και να ανταποκρίνονται καλύτερα στο που χρειάζονται ελάχιστες δεσμεύσεις για την ασφάλεια. Θα πω και δύο λόγια τώρα για την ατζέντα που έχουμε μπροστά μας, το 2015 δηλαδή. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει αρχίσει, πάλι είναι ευάλωτες οι αγορές εργασίας, υπάρχουν πολλές προκλήσεις, προβλήματα με την ανάπτυξη, με τη ζήτηση και υπάρχει απειλή να υπονομευθεί η μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή και στα κατάλληλα προσόντα. Οι αναθεωρήσεις μας έχουν δείξει ότι γίνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να συνεχιστούν αυτές, μερικές φορές να επιταχυνθούν. Πάντως τέτοιες μεταρρυθμίσεις πάντα χρειάζεται χρόνος για να αποδώσουν καρπούς και να ενισχύσουν τις πολιτικές απασχόλησεις. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες αλλαγές μέσα στο 2015. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θα δώσω τώρα στην ε, Πρόεδρο της ε, Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά, αγαπητοί βουλευτές. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα και που σας παρουσιάζω το έργο της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Κάποια πράγματα ως προς το ιστορικό μας. Πρόκειται για μια επιτροπή που δημιουργήθηκε το 2000 βάσει της συνθήκης για την κοινωνική προστασία και περιλαμβάνει και διάφορες ε, τριβές ε, σε τέτοια συζητήματα. Βασιζόμαστε σε δύο πυλώνες, ε, σύμφωνα με αυτά που μας παρουσίασε και προλαλήσαντα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η θεματική εργασία για την ανάπτυξη κοινή συνεννόησης μεταξύ των κρατών μελών για τις προκλήσεις στο κοινωνικό τομέα και να αναζητήσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές. Όπως και οι συναδελφοί λοιπόν ε, σε θέματα απασχόλησης, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας ε, σε ό,τι αφορά το εξάμενα βασιζόμαστε στις εφαρμογή των συστάσεων, στην ε, πολυμερή εποπτεία και η αιτήσια εξέταση της Επιτροπής των Σχετικών Γνωμοδοτήσεων περιλαμβάνει και συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο τελικά αποτελεί και τη βάση των τελικών συστάσεων που εγκρίνει το Συμβούλιο. Η εργασία της ε, Επιτροπής μας και της Επιτροπής Απασχόλησης ε, έχει αποδεχτεί πολύ χρήσιμη, καθότι αποτελεί το μοναδική, η Μοναδική Επιτροπή που εργάζεται ουσιαστικά σε θέματα κοινωνικής ε, συμπερίληψης. Κάνουμε επίσης θεματικές αναθεωρήσεις, εξετάζουμε τις ε, γενικότερες τάσεις ε, σε θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων και την ε, κοινωνική πρόνοια, της συντάξει και το καθεξής. Το 2014 εγκρίναμε δύο σημαντικές εκθέσεις για την σωστή κοινωνική προστασία για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες στην γυράσκουσα κοινωνία και κατά δεύτερον τα κοινωνικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα χρηματοδοτηθεί η αποτελεσματικότητα των, της χρήσης των πόρων. Σήμερα, ε, φέτος θα, θα ολοκληρώσουμε την έκθεσή μας μέχρι το τέλη Μαΐου και έτσι θα κοιτάξουμε κατά πόσο είναι σωστά τα συστήματα ε, συνταξιοδότηση σε ό,τι αφορά και τις ανάγκες της γυράσκουσας κοινωνίας. Θα δούμε και κατά πόσο είναι βιώσιμα τα συστήματα συνταξιοδότησης. Το SPC επίσης ε, καταρτίζει δύο τις εκθέσεις ε, για το Συμβούλιο, καταρχάς σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία και προτάσεις του χρόνου προς το Συμβούλιο για τα ζητήματα αυτά και αυτά ελπίζουμε ότι θα περάσουν στην γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την ε, έρευνά της εκπρόοδου και Ύστερα η δεύτερη έκθεση έχει να κάνει με την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντα υπόψη και, λαμβάνοντας υπόψη και τους δείκτες ε, κοινωνικής παρακολούθησης. Το 2014 ήταν πάρα πολύ σημαντικό έτος για τις εργασίες μας και για το Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά και τη συνεργασία μας με την ΕΜΚΟ, σε ό,τι αφορά την διάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για το 2020 και το ποιος είναι ο τρόπος να έχουμε πιο πολύ κοινωνική Ευρώπη. Από κοινού με την έκθεσή μας με την ΕΜΚΟ αντιμετωπίσαμε και κοιτάξαμε τα θέματα. Ε, μία από τις βασικές προκλήσεις στην έκθεση ήταν η ανάγκη για πιο ισόρροπη διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και λόγω της, ε, του κατεπήγοντος χαρακτήρα της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν βασικά εστιασμένη στις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές της, ε, των κρατών. Σήμερα θεωρούμε ότι έχουν, έχει αγνοηθεί η κοινωνική πολιτική και έτσι λοιπόν ε, βρήκαμε τρεις προτεραιότητες κοινέ ε, στην στρατηγική του 2020 και πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμπερίληψη. Και το πιο σημαντικό είναι επίσης να υπάρχει εθνική δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αυτά. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις στόχους της στρατηγικής, αλλά το πώς θα τους πετύχουμε, η Ευρώπη 2020 και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχουν καταδείξει και αποδείξει την αξία τους ως καταλήτης για μεταρρυθμίσεις. Η εστίαση θα πρέπει να γίνει στην εφαρμογή πλέον των συμπεμφωνημένων μεταρρυθμίσεων που παίρνουν χρόνο και στην συνεχιζόμενη δέσμευση για την εφαρμογή τους, όπου υπάρχει ανάγκη. Μία από τις βασικές βελτιώσεις που υποστηρίζει το Συμβούλιο είναι η βελτίωση της κοινωνικής διακυβέρνησης, πάντα με σεβασμό της επικουρικότητας και της δικαιοδοσία των κρατών μελών και σύμφωνα και με τους στόχους που έχει θέσει η συνθήκη για την κοινωνική προστασία. Χρειαζόμαστε ένα ισόρροπο ευρωπαϊκό εξάμεινο σε ό,τι αφορά και του ενωπημένου στόχους τη στρατηγικής 2020 που θεωρούν ότι είναι βασικός πυλώνας ε, ε, η κοινωνική συμπερίληψη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει εταιρική σχέση μεταξύ των προπροσκευαστικών σωμάτων, της Επιτροπής μας και της ΕΜΚΟ για να ε, βελτιωθούν τα ζητήματα της μακροπρόθεσμης ε, πρόνοιας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον, την έγκριση του πεδίου εφαρμογή τη Επιτροπή μα και τη Επιτροπή ΕΠΚΟ ήταν ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Πρόκειται για ένα εργαλείο μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι επιτροπέ λοιπόν έχουν δεσμευτεί για το scoreboard αυτό ω ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία. Επίση, έχουμε και μια ενοποιημένη προσέγγιση από την, ε, με το πακέτο ε, οικονομικής ε, συμπερίληψης και αποτελεί μία δέσμευση της Νέας Επιτροπής σε ό,τι αφορά το τριπλό α για την Ευρώπη. Αυτή τη δέσμευση την παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και την αποδεχόμαστε και την προσυπογράφουμε και εμείς. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ανάπτυξη και συμπερίληψη, θα πρέπει να γίνουν μακροοικονομικές αλλαγές που θα λαμβάνουν πιο πολύ ε, υπόψη του κοινωνικό αντίκτυπο των επιλογών που γίνονται και αυτό κυρίως λόγω των οικονομικών ωφέλων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι αφορά το πακέτο EGS, η Ευρωνέα Επιτροπή έχει εκφράσει την πρόθεση να ενταχθούν όλα αυτά στο πλαίσιο του συντονισμού για την οικονομική πολιτική. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο στόχος. Αλλά επίσης πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει ενεποιημένη προσέγγιση στο HSP1, όπου θα δίνεται εξίσου έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη με τα σωστά εργαλεία και μάλιστα και στα σωστά φόρα. Κλείνοντας, τρία μηνύματα θα ήθελα να σας διαβιβάσω σήμερα στο πλαίσιο της νέας επιτροπής και της και επενδυτικής ατζέντα. Οι επενδύσεις σε θέματα κοινωνικά θα πρέπει να παίζουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Και σε ό,τι αφορά την οικονομική απόδοση, πάντα θα πρέπει να υπάρχει συμπεριλήψη του κοινωνικού αντικτύπου. Αν θέλουμε να υπάρχει συμπεριλήψη σε ό,τι αφορά την οικονομική ατζέντα, θα πρέπει να θέσουμε στόχους κοινωνικούς και να είμαστε πολύ δεσμευμένοι σε ό,τι αφορά τους στόχους και τις στρατηγικές που εφαρμόζουμε. Και τέλος, θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόμο που παρακολουθούμε την κοινωνική ανάπτυξη και να δίδεται ίση προσοχή και σε αυτούς τους παράγοντες όπως και στην οικονομική ανάπτυξη. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια μιας ενοποιημένης πολιτικής που θα δίνει ε, έμφαση σε όλους αυτούς τους φορείς και στις αρμόδιες ε, ε, αποφάσεις, τις ε, ανάλογες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την εισαγωγή της σας. Ε, we'll go to the, ε, Περνάμε στους συντονιστές που μπορούν να θέσουν ερωτήσεις. Από ε, το ΕΛΚ, κυρία Μωρά Ζαπιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την παρουσίαση που κάνατε και τους δύο πρόεδρους για τις δύο παρουσιάσεις. Ήταν πολύ διαφωτιστικές. Μετά από τις παρουσιάσεις έχω κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Μπέβερς καταρχήν. Τονίσατε ότι μελετάτε την ανεργία των νέων. Ε, μελετάτε και την ε, εγγύηση για την νεολαία. Παράλληλα, μελετήσατε την εφαρμογή της ε, εγγύησης ε, για την νεολαία και την πρωτοβουλία για τους νέους. Δύο πολιτικές που είναι πολύ κοντά. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι η ενίσχυση της εγγύησης για την νεολαία στις ε, πιο δύσκολες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θέτω αυτό το ερώτημα είναι γιατί βλέπω πολλή σύγχυση σε όλα τα πολιτικά επίπεδα και είναι δραματικό που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θέλουν να κάνουν ε, επικοινωνιακή πολιτική με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ε, ενώ αυτό που κατάφεραν είναι να προκαλέσουν σύγχυση στο μυαλό όλων. Τελικά, τι συμβαίνει. Δεύτερον, εδώ δώσαμε μάχη σε αυτή την Επιτροπή για να πάει το 20% του κοινωνικού ταμείου για την καταπολέμηση της στόχιας μέσω της κοινωνικής ένταξης. Τι αποτελέσματα έχετε για το θέμα αυτό. Και τρίτο ερώτημα. Χρειάστηκε επίσης να δοθεί μάχη, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να μην ενσωματωθεί στο Ταμείο Συνοχής. Ποια είναι η θεώρησή σας, ποιο είναι το όραμά σας για την χρήση των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου και για το πώς εφαρμόζονται τα κονδύλια. κυρίως να μου μιλήσετε δηλαδή για τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από αυτό και την εφαρμογή τους. Τρίτον, η εξέλιξη προς τις αρμοδιότητες. Μιλήσαμε πολύ για την επικύρωση της επαγγελματικής εμπειρίας και των δεξιοτήτων. Επί 15 χρόνια τα λέμε αυτά. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν πάει καλά. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να κάνουμε, ούτω ώστε να ενθαρρύνουμε πραγματικά τους μισθωτούς με ας πούμε μακριά καριέρα ε, τη δυνατότητα επικύρωσης των αδεξιοτήτων τους. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Γιούτα Στάιν από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Στανιρούκο που είσαστε εδώ μαζί, σήμερα, μαζί μας σήμερα και για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και κυρία Μαρανσάτια ανέφερε το πιο σημαντικό θέμα για μας, την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Αλλά, από την άλλη, υπάρχει και μία ολοένα και αυξανόμενη μακροπρόθεσμη ανεργία στην Ευρώπη. Τι μέτρα λοιπόν θεωρείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στοχευμένα εδώ στην Ευρώπη. Προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροή σε αυτούς τους κόσμους οι οποίοι ε, μακροπρόθεσμα χάνονται από την αργόρα εργασίας και από την κοινωνία όμως. Η πολιτική λιτότητα στην Ευρώπη έχει καταστρέψει πολλά πράγματα. Χρειάζομαστε κατεπηγόντως επενδύσεις. Κύριε Ντομινίκ, είπατε ότι το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει κατεπηγόντως να περιλαμβάνει και κοινωνικούς στόχους, κοινωνικές πτυχές. Πού θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν αλλαγές σε σχέση με αυτά που μας παρουσίασε εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα έπρεπε να σημειωθεί βελτίωση. Κύριε Ντομινίκ, μιλήσατε για τις συντάξεις, για τη γύρανση της κοινωνίας και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή. Έχετε κάτι συγκεκριμένο να προτείνετε, έχετε κάποια συγκεκριμένη ιδέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι την τελευταία εβδομάδα δημοσίευσε την ε, ετήσια έκθεση για τους κοινωνικούς ε, στόχους και στην πρώτη ανακοίνωση τύπου η Κομισιόν είπε ότι θα πρέπει οι χώρες να έχουν καλές θέσεις απασχόλησης, καλή προστασία και ανθρώπινες ε, συνθήκες εργασίας και τότε θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κρίση. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί λοιπόν δεν ε, έχουν κάνει βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κάρη από την oh, GUNGL. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές για τα εισαγωγικά του σχόλια τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τη δουλειά σας. Μιλήσατε και οι δύο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι τμήμα της οικονομικής διακυβέρνησης των κρατών μελών αυτό. Θα πρέπει να δούμε τη δομή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι κάτι το οποίο το συζητάει η Κομισιόν, εμείς το συζητάμε. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι το πώς λειτουργεί η οικονομική διακυβέρνηση. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Οι κοινωνικές παράμετροι και οι κοινωνικοί δείχτες θα πρέπει να ενσωματωθούν ενδεχομένως στο εξάμεινο αυτό, ούτως ώστε να μετράμε την, το επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Οι μεγάλες οικονομικές παράμετροι, όπως το δημοσιονομικό έλλειμμα, μοιάζει να είναι ο πιο βασικός δείχτης ή το χρέος, ας πούμε, είναι η πιο βασική δείκτε αυτή τη στιγμή του εξαμήνου. Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη μα την απασχόληση και την κοινωνική προστασία, ούτω ώστε να μην είναι υποδέστερο σε σχέση με τους οικονομικούς ε, δείκτε. Γιατί χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε θέσεις ε, απασχόλησης. Τι διαφορετικές αλλαγές πρέπει να κάνουμε για να σωματώσουμε αυτό το στοιχείο. Η Λάουρα Ατζέα από την EFTD. Ε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που μας κάνατε και τους δύο. Χρειαζόμαστε ίσως και, άλλους, και άλλα στοιχεία και άλλους δείκτες. Δύο ερωτήσεις και δύο αξιολογήσεις σε σχέση με την κατάσταση ε, στην Ιταλία της εγγύησης για την νεολαία. Μέχρι σήμερα έχει αποτύχει δεν υλοποίησε τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν υπάρχει ούτε πρόσβαση ούτε επικοινωνία γύρω από αυτό. Διερωτώ με το λάθος είναι στον τρόπο που εφαρμόζεται ή υπάρχει έλλειψη συντονισμού επίσης. Συντονισμός που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μεταξύ αυτών που τον συλλαμβάνουν ως ιδέα και αυτών που το εφαρμόζουν. Γιατί σε ορισμένε χώρε που εφαρμόστηκε ήταν αποτελεσματικό και έδωσε πολύ θετικά αποτελέσματα. Αλλά μέχρι στιγμή στην Ιταλία είναι ένα project το οποίο δεν χρησιμοποιείται, χάθηκε στους μεάνδρους της γραφειοκρατίας και οι νέοι εκ των προτέρων δηλαδή σιγά μην το χρησιμοποιήσω. Επίσης, μιλήσατε για την κοινωνική διάσταση που θα πρέπει να έχει το ίδιο επίπεδο, να εξισορροπείται, να εξισώνεται μάλλον με την μακροοικονομική και οικονομική διάσταση. Μια και μιλάμε μόνο για στόχους ε, εξισορρόπηση του προπολογισμού, για διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, για μη υπέρβαση του ορίου ε, ελλείμματος προς ΑΕΠ. Υπάρχουν κάποιες ε, θέσεις, ας πούμε, των κρατών μελών. Ε, δεν νομίζω ότι η κοινωνική διάσταση είναι στο ίδιο επίπεδο με την οικονομική διάσταση. Έπρεπε να είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά σήμερα η οικονομική διάσταση, οι κανόνες γύρω από αυτήν και τα όρια είναι οι πιο αποφασιστικοί. Οι στόχοι της ε, οικονομικής πολιτικής ε, είναι αυτοί που πρέπει να υλοποιηθούν υποτίθεται και ποιος πληρώνει το τίμημα η κοινωνική διάσταση. Τώρα, για τις ε, συντάξεις, κάποιες πληροφορίες. Το πρόβλημά μας είναι τρομακτικό στην Ιταλία. Έχουμε ελάχιστες συντάξεις, πολύ κάτω από τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης. Έχουμε πρόορη συνταξιοδότηση σε επίπεδα πολύ χαμηλά. Πώ θα μπορούσαν τα πράγματα να αλλάξουν και στο επίπεδο των συντάξεων μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίε. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Μπέβερς. Όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τις ερωτήσεις που μου κάνουν οι ευρωβουλευτές να μιλήσω για την ανεργία, η απασχόληση των νέων και την, το σχήμα εγγύησης για την νεολαία. Στην ΕΜΚΟ παρακολουθούμε την, τον τρόπο εφαρμογής της εγγύησης για την νεολαία εκ του σύνεγγυ. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από δείκτες για να παρακολουθήσουμε ακριβώς το πώς εφαρμόζεται και μέχρι στιγμής ε, κάναμε τρεις αναθεωρήσεις του μέτρου αυτού όπου συζητήσαμε το πώς εφαρμόζεται η εγγύηση για την νεολαία και στα 28 κράτη-μέλη αυτό που βλέπουμε είναι προφανώς μια μεικτή εικόνα, όπως είναι αναμενόμενο. Ορισμένες χώρες είχαν ήδη κάτι που έμοιαζε πολύ με, τις, ε, με την εγγύηση για την νεολαία. Κάποιες άλλες χώρες άρχισαν να τελείως, ξεκίνησαν από τελείως διαφορετική αφετηρία. Επιπλέον, Υπάρχει όντως μια σύγχυση ανάμεσα στην εγγύηση για την νεολαία και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ειδικά για τις χώρες που δεν λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από την πρωτοβουλία για την απασχόληση. Μερικές φορές χρειάστηκε να ασκηθεί μεγαλύτερη πυθός για να εφαρμόσουν και την εγγύηση για την νεολαία οι άλλες χώρες που λαμβάνουν αυτή την οικονομική βοήθεια και πολύ σωστά, ο στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν ότι αυτό που δημιουργούν και ότι οι μεταρρυθμίσεις που κάνουν για να εξασφαλίσουν ότι η εγγύηση για την νεολαία μπορεί να εφαρμοστεί είναι βιώσιμες τη μέρα που θα σταματήσει η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Η εγγύηση για την νεολαία θα πρέπει να θεωρηθεί μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση η οποία βελτιώνει η μετάβαση από το σχολείο στο χρόνο εργασία με βιώσιμο τρόπο. Και η πρωτοβουλία και τα λεφτά που υπάρχουν είναι απλώς ένα μέσο, για να, ένας τρόπος για να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Αλλά ο στόχος ποιος είναι. Ο στόχος είναι η εγγύηση που θα εξακολουθήσει να υπάρχει χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Η εγγύηση των νέων λοιπόν είναι πιο, το πιο διαρκές ας πούμε κομμάτι, το πιο μακρόπνο. Η μεικτή εικόνα αυτή δείχνει ότι σε ορισμένε χώρε έχει σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι σε άλλε. Αλλά έχουν όλες οι χώρες αρχίσει να δημιουργούν εταιρικέ σχέσεις που δεν υπήρχαν πριν. Οι περιφερειακές αρχές συνομιλούν μεταξύ τους, οι φορείς οι εκπαιδευτικοί συζητούν με ιδρύματα της αγοράς εργασίας δημιουργούνται γέφυρες μεταξύ της εκπαίδευσης και της, του χώρου της απασχόλησης. Το γεγονός ότι σε ορισμένε περιπτώσεις δεν βλέπετε απτά και άμεσα αποτελέσματα είναι φυσικό σε χώρες που οι προκλήσεις είναι τρομακτικές. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο πριν δρέψουμε τους πρώτους καρπούς. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι, και ξέρω λιγάκι την Ιταλική περίπτωση, ότι οι δομές που δημιουργούνται, οι εταιρικέ σχέσεις που στείνονται, είναι πραγματικά ένα βήμα προς το εμπρός. Η επικοινωνία για την εγγύηση για την νεολαία είναι σε, στα σπάργανα σε πολλές χώρες και θα μπορούσαν να γίνουν διάφορα πράγματα για να γνωρίσουν οι νέοι τις δυνατότητε που υπάρχουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εμείς δεν εμπλεκόμαστε τόσο, όχι άμεσα τουλάχιστον, όμως προφανώς συνδέεται προφανώς το Ταμείο αυτό με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για το πώς οι χώρες θα χρησιμοποιήσουν τα, με, τα μέσα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ελπίζουμε να επικεντρωθούν στις βασικές προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί στο εξάμεινο. Η μακροχρόνια ανεργία τώρα και η επικύρωση των δεξιοτήτων. Αυτά συνδέονται για μένα άρρηκτα. Ένας από τους βασικούς στόχους που έχουμε είναι να καταπολεμήσουμε την μακροχρόνια ανεργία με τα δικά μας μέσα. Φυσικά αυτό θα γίνει και μέσω της οικονομικής ανάπτυξης. Ε, της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι κοινωνικές πτυχές για μας είναι σημαντικές, όπως ενεργές πολιτικές για την ε, αγορά εργασίας. Ε, ετοιμοπαράδοτη βοήθεια, ας πούμε, η βοήθεια που χρειάζεται ο καθένας στα μέτρα του κομμένη. Δεν ξεκινάνε όλοι μακροχρόνια άνεργοι. Από την αρχή θα πρέπει να, με το που θα μείνουν άνεργοι θα πρέπει να τους ε, βάλουμε ξανά στην αγορά εργασίας. Ε, ορισμένες ε, χώρες έχουν ενδιαφέροντα συστήματα profiling, ούτω ώστε πολύ νωρίς να βλέπουν ποιοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι να γίνουν μακροχρόνια άνεργοι και να το αντιμετωπίσουν πάρα αυτά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα καλά παραδείγματα που έχουμε για να πείσουμε και άλλες χώρες ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα. Για το εξάμεινο, για την εξισορρόπηση που πρέπει να κάνουμε, για το αν θα πρέπει να κάνουμε αλλαγέ στη δομή. Δεν νομίζω ότι η μηχανική, η λειτουργία του εξαμήνου είναι μη ισορροπημένη και πρέπει να αλλάξει. Το σύστημα το οποίο υπάρχει, νομίζω, καταρχήν επιτρέπει μια εξισορρόπηση των ε, κοινωνικών και οικονομικών μελημάτων. Φυσικά οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται μέσω του εξαμήνου είναι αυτές που πρέπει να εξισορροπηθούν και οι πολιτικές επιλογές που γίνονται στα πλαίσια του εξαμήνου θα πρέπει να εξισορροπηθούν. Και μια και μοιάζει ας πούμε να βγαίνουμε λιγάκι δειλά-δειλά από την κρίση, Μέσω του εξαμήνου μπορούμε να κάνουμε πολιτικές επιλογές ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι πως οι δύο διαστάσει κοινωνική και οικονομική είναι ισορροπημένε. Φυσικά υπάρχει και σχέση με τους δείκτε που χρησιμοποιούνται. Ένα στοιχείο του εξαμήνου είναι η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Στο δικό μας σύστημα δικτών έχουμε το πίνακα αποτελεσμάτων για τα κοινωνικά θέματα και την απασχόληση. Και όπως είπε θα πρέπει να δημιουργήσουμε πιο έντονε σχέσεις ανάμεσα στα δύο συστήματα των μακροοικονομικών ισορροπιών και του το πίνακα αποτελεσμάτων, ώστε να μην θεωρούνται τόσο κόσμοι, ας πούμε. Και θα πρέπει μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συνέχεια να έχουμε ολοκληρωμένε πολιτικές με την κοινωνική και την οικονομική διάσταση. Ευχαριστώ πολύ από τα διάφορα που άκουσα είναι το πακέτο το επενδυτικό της Επιτροπής και πώς θα χρησιμοποιηθεί ως κοινωνική επένδυση. Αυτό έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά προβλήματα. Έχουμε τη μακροχρόνια ανεργία και εδώ είναι που συγκεντρώνονται όλα. Τα κοινωνικά συστήματα, όπως τα έχουμε σήμερα, πρέπει να προσαρμοστούν, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να επενδύσουν τα κοινωνικά συστήματα και να δώσουν πόρους στα συστήματα αυτά ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά μας. Για τη μακροχρόνια ενεργεία πιο συγκεκριμένα έχετε προγράμματα που προσαρμόζονται στο γεγονός ότι γερνάει το εργατικό δυναμικό. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη ελαστικότητα, να επιτρέπουμε να μπορούν προσωπικά να προσαρμόζονται οι άνθρωποι και να παραμένουν στην αγορά εργασίας αντί να φεύγουν και να μένουν ε, άνεργοι. Αυτές τις προσεγγίσεις εξετάζουμε. Και βέβαια θέλουμε την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα συζητηθεί στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες παραμέτρους. Έχουμε συζητήσει για τις συντάξεις επίσης. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι το εργατικό δυναμικό πρέπει να προσαρμοστεί σε περισσότερα χρόνια δουλειάς, εφόσον ζούμε και περισσότερο. Αλλά πρέπει να οργανώνεται το εργατικό δυναμικό από μόνο του για να υπάρχει προσαρμογή και των κοινωνικών συστημάτων σε αυτά. Άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές για να αντιμετωπίσουμε και να προσαρμοστούμε στις δημογραφικές αλλαγές. Αυτό σημαίνει εξυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Συγχρόνως με τις συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σεβόμαστε κάποιες κοινωνικές αρχές και αξίες που έχουμε στην Ευρώπη. Που είναι σημαντικό και αυτό και εδώ είναι που έρχομαι σε ελάχιστε ε, συντάξεις που είπατε για την Ιταλία. Πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Να ελέγχουμε το επίπεδο των ε, επιδομάτων που δίνουμε στους πολίτες. Να υπάρχει κάποιο κριτήριο για να ξέρουμε τι μέτρα κοινωνικής πολιτικής μπορούμε να υιοθετήσουμε για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς οι πολίτες. Για αυτές τις κοινέ κοινωνικές αξίες πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο στο μέλλον. Θα είναι ένας ε, από τους κύριους στόχους μας, ε, τα κύρια θέματα που θα έχουμε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής μας. Τέλος, για την κοινωνική διάσταση πώς συνδέονται τα κοινωνικά ζητήματα με το εξάμεινο, όπως είπε και ο συνάδελφος, έχουμε τα εργαλεία γι' αυτό. 2013 είχαμε μία σε βάθος συζήτηση για την απασχόληση και το κοινωνικό βαθμολόγιο, τον πίνακα επιδόσεων. Είναι ένα καλό σημείο κίνησης αυτό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα λοιπόν από την Επιτροπή είναι το κοινωνικό στοιχείο να συμπεριληφθεί περισσότερο στις μακροοικονομικές εκτιμήσεις. Και συνεργαζόμαστε και με τους άλλους εταίρους. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και σίγουρα σύντομα θα υπάρξουν συζητήσεις στις επιτροπές μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βακενισούτε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο καλεσμένους μας, και τον κύριο Μπέβερς και τον κύριο Ντομινίκ, που μας παρουσίασαν το έργο των επιτροπών τους. Θέλω να ρωτήσω τα Και οι δύο επιτροπές εκπονούν συστάσεις, η καθεμία στον τομέα της, για κατευθυντήριες γραμμές στην απασχόληση, για την αναθεώρηση των συστημάτων κοινωνικής ε, προστασίας, συστάσεις προς τις χώρες. Η ερώτησή μου είναι, δεδομένου ότι εργάζεστε πολύ εντατικά, οι χώρες μέλη έχουν την πολιτική βούληση να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις που τους κάνετε ώστε να επηρεαστεί έτσι η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Μπέβερς είπε ότι ίσως χρειαζόμαστε κάποιες ε, υποχρεωτικές δεσμεύσεις, δηλαδή όχι μόνο κατευθυντήριες γραμμές, αλλά υποχρεωτικά μέτρα που θα έπρεπε να υιοθετήσουν οι χώρες μέλη βάσει των ευρημάτων σας. Για παράδειγμα, για την ε, εγγύηση για τους νέους. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι δεσμευτικό, υποχρεωτικό. Η άλλη μου ερώτηση είναι, οι επιτροπές σας έχουν συζητήσει ποτέ ή σχεδιάζετε να συζητήσετε τις επιπτώσεις της μετανάστευσης. Εγώ πολύ χαίρομαι που έχουμε την ελευθερία κυκλοφορίας, όμως μερικές χώρες χάνουν τον πληθυσμό τους διότι ο κόσμος φεύγει, η μετανάστευση δηλαδή από την Ευρώπη ή από τις ευρωπαϊκές μερικες χωρες χανουν τον πληθυσμο τους διοτι ο κοσμος φευγει αλλού από την γυραιά Ευρώπη φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες υπήρους. Σκοπεύετε λοιπόν να ασχοληθείτε καθόλου με αυτό το φαινόμενο. Να κάνετε κάποια έρευνα που να είναι χρήσιμη για τις χώρες μέλη. Πιστεύω ότι το κοινωνικό μοντέλο πια είναι μια ωραία ανάμνηση. Με την τεράστια ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ένδια, είναι πράγματα τα οποία αυξάνονται αντί να μειώνονται. Ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν, οι επιτροπές σας θα μπορούσαν να καταλήξουν σε προτάσεις εγγύηση για τα παιδιά για παράδειγμα. Έχουμε τόσο μεγάλο επίπεδο φτώχειας για τα παιδιά, όλους μας πονάει. Εντάξει, έχουμε την εγγύηση για τους νέους, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τις ρίζες, τη βάση τα παιδιά μας που ζουν σε φτώχεια από τότε που γεννιούνται. Καταλαβαίνετε ότι όταν θα γίνουν νέοι δεν έχουν πια τα κίνητρα να δουλέψουν, να κερδίσουν χρήματα και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Να πάμε λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα της φτώχειας των παιδιών, των μικρών παιδιών. Πώς είναι δυνατόν να ζούμε στην πλουσιότερη ήπειρο στον κόσμο και να εξακολουθούμε να έχουμε φτώχεια στα παιδιά. Θα ήθελα συστάσεις από αυτόν παρακαλώ. Ευχαριστούμε κυρία Αλάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας για τις παρουσιάσεις σας. Κύριε Μπέβερς, δεν συμμεριζόμαστε καθόλου την αισιοδοξία σας, για κανένα σημείο θα έλεγα και κυρίως όταν λέτε πως βλέπετε να απομακρύνεται η κρίση. Εμείς πιστεύουμε ότι το αντίθετο ισχύει και ότι είναι πολιτική ευθύνη, ακόμα και αν βλέπουμε κάποιες αυθύνες φωτός, φοβάμαι ότι πάμε προς τα χειρότερα. Το κοινωνικό σύστημα χρηματοδοτείται από τον εθνικό πλούτο ως επιτοπλίστων. Η Ευρώπη δυσκολεύεται να βάλει τάξη στα οικονομικά της. Όλες οι χώρες έχουν τεράστιο χρέος. Και δεν είναι η σημερινή δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα αλλάξει τα πράγματα. Η χρηματοδότηση γίνεται επίσης από την εργασία. Όμως αυτήν την Επιτροπή ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο χαμηλή είναι απασχόληση και ποιοτικά και ποσοτικά. Είναι πήγον λοιπόν κατά τη γνώμη μας να κάνετε προτάσεις που να αλλάξουν την κατάσταση, να είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Μέτρα δυνατά και μέτρα αλλαγής και όχι να προσαρμοζόμαστε στα παλιότερα μέτρα τα οποία αποδείχθηκαν τόσο ελληματικά. Και για σας κύριε Ντομινίκ δεν συμφωνώ με την ιδέα σας για τον εξυγχρονισμό. Αν εξυγχρονισμός είναι να δουλεύουμε πιο πολύ, ε, εντάξει μπορεί να έχω και ίδιο συμφέρον βέβαια που το λέω, αλλά τι θα συμβεί. Η συνταξιούχοι θα διακόπτουν την εργασία τους κάθε φορά που είναι άρρωστοι και θα διακόπτουν κάποια στιγμή γιατί δεν θα τους το επιτρέπει η υγεία τους. Και έτσι κι αλλιώς η πρόοδος της ε, κοινωνίας μας θα πρέπει να είναι καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας όσο και κατά τη διάρκεια της σύνταξης. Δεν μπορεί νεκρός μόνο να παίρνει τη σύνταξή του κάποιος. Πρέπει λοιπόν έγκαιρα να φροντίσουμε να παίρνουμε και τη σύνταξή μας για να μπορούμε να υποφελούμαστε και από αυτήν. Ευχαριστούμε κύριε Πάλλας. Ευχαριστώ και τους δυο σας για τις παρουσιάσεις σας. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, μελετήθηκε καθόλου από τις επιτροπές σας η περίπτωση ενός συστήματος ανεργία σε περίπτωση ασύμετρου σοκ, όχι μόνιμα, έτσι, ε, από κοινού του συστήματος ταξιδοτήσεων, κάπως όπως έχει το αμερικανικό σύστημα, για να κάνω αυτή τη σύγκριση. Δεύτερον, ερώτηση και παρατήρηση. Μια που το προσδόκιμο ζωής αυξάνει, πρέπει να δουλεύουμε και περισσότερο, έτσι λέμε. Άρα να παίρνουμε αργότερα σύνταξη. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το εξή. Εξαιτία τη ανεργία, εξαιτία τη μερική απασχόληση, εξαιτία του γεγονότο ότι οι άνθρωποι δεν δουλεύουν ε, επί μόνιμη βάση, αλλά υπάρχουν περίοδοι όπου δεν δουλεύουν και κάποιοι δεν θέλουν εργαζόμενους πάνω από 50 ετών, τελικά στα 58 στη Γαλλία δεν μπορεί να δουλέψει πια κανείς. Και αν αυξήσουμε τον ε, χρόνο πρέπει να δουλεύει κανείς, αυτό που θα αναγκαστούμε να κάνουμε θα είναι να μειώσουμε τις συντάξεις. Λέμε ζούμε περισσότερο, άρα πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο. Μα δεν φτάνει, πρέπει να είναι εφικτό αυτό. Και να αναρωτηθούμε επίσης και γιατί υπάρχει ανεργία. Λείπει η ανάπτυξη μόνο ή η παραγωγικότητα αυξάνει με την ψηφιοποίηση ή με την μηχανική και τελικά δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που παράγουν. Και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Ωραία, απαντήσεις τώρα, κύριος Μπέβερ πρώτα. Ευχαριστώ για τις ειδικέ αναχώρες συστάσεις καταρχάς. Και ποια είναι η φύση τους. Στην τελική συστάσεις είναι. Εμείς ως Επιτροπή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι ότι έχουν νόημα, ότι είναι προσαρμοσμένες ανάγκες, πολιτικά ρεαλιστικές και προσπαθούμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου να πιέσουμε σοβαρά τις χώρες, ούτως ώστε να παρακολουθήσουν το πρόβλημά τους, ούτως ώστε να αξιοποιήσουν όσο μπορούν τις συστάσεις, όμως την τελική πολιτική ευθύνη την έχουν και πρέπει να την έχουν τα κράτη-μέλη. Είναι δική τους ευθύνη τελικά να χρησιμοποιήσουν αυτές τις συστάσεις ως πολιτικά εργαλεία, εργαλεία πολιτικής. Η φύση της διαδικασίας είναι δεδομένη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε καλές συμβουλές στις χώρες. Υπάρχουν και τρόποι να ασκήσουμε πίεση στις χώρες. Όμως την πολιτική ευθύνη τη φέρουν οι χώρες και μόνο αυτές. Για την μετανάστευση και τις διάφορες πτυχές της μετανάστευσης. Αν δείτε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μέχρι στιγμής, η διατύπωση είναι αρκετά αόριστη, υπάρχει πολλή αοριστολογία. Συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να συζητήσουμε πιο ενδελεχώς το θέμα και ετοιμάζουμε το πρόγραμμα εργασίας ε, του 2015 ε, και εντός αυτού σκοπεύουμε να συζητήσουμε την οικονομική μετανάστευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε κάποιες συμβουλές πολιτικής ε, με περισσότερη, περισσότερο ζουμί, ας πούμε, παρά τις γενικολογίες που είχαμε μέχρι τώρα. Πέρυσι, κάναμε μια συζήτηση όντως για τη δυνατότητα κάποιου μηχανισμού επιδομάτων ε, ανεργίας. Κοινό πανευρωπαϊκό ή στην ΟΝΕ. Ήταν μια γενική θεωρητική συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία πραγματική πρόταση πολιτικής φύσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν. Σκεφτήκαμε απλώς ότι θα ήταν χρήσιμο εμείς ως Επιτροπή που είμαστε εξοικειωμένοι με το πώς λειτουργούν τα επιδόματα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Δεν καταλήξαμε σε μονοσήμαντα συμπεράσματα όμως, όμως παρουσιάσαμε μία σύντομη έκθεση στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Και κυρίως τι είπαμε, ποια είναι τα διαφορετικά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ε, μηχανισμούς επιδομάτων, ας πούμε, ανεργίας. Ένα πανευρωπαϊκό μηχανισμό, ας πούμε, μην ξεχνάτε ότι τα σημερινά συστήματα είναι ποικίλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι τεχνικές περιπλοκές όλων των μοντέλων που προτείνονται δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Φυσικά η τελική απόφαση δεν είναι τεχνική, είναι πολιτική. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και την τις τεχνικές περιπλοκές. Τώρα, υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν μια αγορά εργασίας ανοιχτή σε όλες ε, τις ηλικίε εργαζομένων. Γίνεται αυτό, απλώς χρειάζονται αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και οι εργοδότες, αλλά και οι δημόσιοι φορείς εξέβρεσης εργασίας μερικές φορές δεν ε, επενδύουν σε πιο ηλικιωμένους εργαζόμενου. Γιατί δεν είναι πεπισμένε αυτά τα όργανα, αυτοί οι φορείς, ότι μπορούν να βρουν δουλειά. Πρέπει να δούμε το πώ λειτουργεί συνολικά η αγορά εργασία μα. Και συμφωνώ ότι το θέμα δεν είναι να πούμε ότι α, κανείς θα παίρνει σύνταξη πιο γέρο ας πούμε, πιο αργά. Πρέπει να, γίνει, να υπάρξει δράση και εντό τη αγορά εργασία. Αλλά ευτυχώ βλέπουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλου του εργαζόμενου. και αυτό είναι σημαντικό και είναι σημαντική και η δουλειά που κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση η Επιτροπή μας, γιατί επιτρέπει στα κράτη-μέλη να μάθουν το ένα από το άλλο και μην ξεχνάμε εξάλλου ότι σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κοινέ προκλήσεις, πολλές κοινέ προκλήσεις. Ο κύριος Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Ε, ακούσαμε διάφορα ζητήματα, αλλά η λογική είναι πάντα σχετική και στο ίδιο πνεύμα. Ποιο είναι ο κοινωνικό αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ποιο είναι ο κοινωνικό αντίκτυπος λοιπόν ε, των μέτρων που λαμβάνονται στα κρατημέλη. Αυτή η συζήτηση για το μεγαλύτερο όριο ηλικία συνταξιδοτότησης είναι πολύ ενδεικτική. Θα πρέπει να δούμε τα συστήματά μα. Αν θέλουμε ο κόσμο να εργάζεται πιο πολύ. Αν θέλουμε καταστάσεις όπου θα υπάρχει λύση για τη δημογραφική αλλαγή. Αυτή είναι άλλωστε και η επιχειρηματολογία για να παραμένει ο κόσμος πιο πολύ στην αγορά εργασίας, πρέπει να προσαρμόσουμε το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίζουμε ότι δεν τιμωρούμε τον κόσμο όταν εργάζεται πιο πολύ. Θα πρέπει να είναι σωστό το ύψος των επιδομάτων. Αυτό θα γίνει λοιπόν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, εξυγχρονίζοντας τα σύγχρονα σταξιδιωτικά συστήματα. Θα πρέπει να αποτεχτούμε ότι ενδεχομένω θα έχουν πιο πολλά προβλήματα υγεία. Θα πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν νέα ε, συστήματα κοινωνική ασφάλεια για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι νέε καταστάσει. Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για εξυγχρονισμό των ε, συστημάτων κοινωνική προστασίας. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην κοινωνική προστασία, αυτό εννοείται. Επανέρχομαι στο θέμα της φτώχεια, της φτώχεια των παιδιών. Υπάρχει φτώχεια μεταξύ των παιδιών στην Ευρώπη. Το πρόβλημα στο σημείο αυτό είναι ότι θα πρέπει να μην αναπαράγεται αυτή η φτώχεια. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Ε, είμαστε λοιπόν στην μέθοδο ανοιχτής, ανοιχτού συντονισμού. Μιλάμε για ήπιο δίκαιο και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι πολλή δουλειά έχει γίνει για την ε, ε, φτώχεια των παιδιών σε ό,τι αφορά τις συστάσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να αποτευχθεί αυτό στο μέλλον. Πολλά λοιπόν έχουν γίνει και το έργο αυτό θα πρέπει να προβληθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ενδεχομένω να τεθούν κάποιες τιμές αναφοράς για να δούμε κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις συνάδουν με τις κοινέ συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στις αρχές που έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ και μια τελευταία ερώτηση πρωτού ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες από τον κύριο Λόπες. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Μια συγκεκριμένη ερώτηση παρακαλώ για μια σύσταση περσινή της Επιτροπής που είχε να κάνει με την ε, επιχειρηματική αποτυχία. Δεν μπόρεσαν ε, να την εφαρμόσουν οι χώρες μέλη. Ξέρω ότι μετά από 18 μήνες έπρεπε να γίνει έτσι μια αναθεώρηση. Εγκρίθηκε τον Μάρτιο που μας πέρασε ήταν μια σύσταση που έλεγε ότι έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την αναδιάρθρωση χρεών και κίνηση των επιχειρήσεων, προκειμένου να δοθούν έτσι κίνητρα και επιχειρηματικά σχέδια. Θέλω λοιπόν να μάθω τι πληροφορίες έχετε για την εφαρμογή που έγινε από τα κράτα μέλη της σύσταση αυτής και πώς ενθαρρύνετε εσείς ε, τα κράτη να εφαρμόσουν τις συστάσεις. Και τι γίνεται με τα άτομα, γιατί καλά οι επιχειρήσεις, δεν θα έπρεπε το ίδιο να το κάνουμε και για τους ανθρώπους. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν ε, ε, νομοθεσίες όταν πρόκειται για πτώχευση μιας επιχείρησης, υπάρχουν συστάσεις από διάφορους διεθνείς οργανισμούς κτλ. για να υπάρχουν συγκεκριμένα στάνταρτ προδιαγραφές. Η Γαλλία για παράδειγμα, έχει ένα νόμο που εφαρμόστηκε σε 150.000 για ατομική πτώχευση. 100.000 στη Γερμανία. Στην Ισπανία κάτω από 1.000 ήταν αυτοί που αποφελήθηκαν. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά η Ισπανία έχει τεράστιο πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι χάνουν το σπίτι τους, τους παίρνουν το σπίτι, έχουν υποθήκη, δεν μπορούν να πληρώσουν και τους το παίρνουν το σπίτι. Με την κρίση είχαμε 400.000 τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που τους βγάλαν από το σπίτι τους. Φοβερές περιπτώσεις και τελικά δεν μπορούν καν να πάρουν τα σπίτια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, παρά τα πολύ χαμηλά επιτόκια που ήταν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η σύσταση υπάρχει. Να δούμε πώς μπορούμε λοιπόν να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι ο θάνατος των ε, πολιτών με τη διάστασή τους, τη διάσταση του πολίτη δηλαδή, εξαιτία των πολιτικών που ακολουθούμε. Ο κύριος Μπέβερς. Α, ο κύριος Δομινίκ. Ναι. Αυτό είναι το τοπινγκ της κοινωνικής στόχιας. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό γενικά. Αν εξετάσουμε το θέμα αυτό με τις υποθήκες και τα σπίτια, όντως είναι ένα δείγμα της στόχιας που παρατηρούμε. Είναι λοιπόν ένα από τα θέματα τα οποία καλύπτουμε εμείς στην ανάλυση μας, στην Επιτροπή μας. Αλλά συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, προκειμένου να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες συστάσεις με την έννοια του να δώσουμε τις καλύτερες δυνατόν λύσεις για να αποφεύγονται ακριβώς αυτές οι περιπτώσεις όσων στις οποίες αναφερθήκατε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο λοιπόν που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ήταν πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή αυτή απόψεων. Ελπίζω να μας ξανάρθετε. Σε λίγα λεπτά, στις 10 και 4 ακριβώς, θα αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Okay, we'll Να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Ταμείο Προσαρμογή στην ε, ε, ε, Παγκοσμιοποίηση, έγκριση νομοδότηση, υπομορφή επιστολή, ε, έναξη ψηφοφορία. Ευχαριστώ, πέρας. Περισσεύει μία ψήφος από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Πέρα ψηφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερη επιστολή σε ό,τι αφορά το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Κέιτερ Πίλερ, υπέρ. Μάλλον έναξη ψηφοφορίας η πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτη περίπτωση για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μίταλ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπέρ. Και τώρα περνάμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συμβιβασμό 1. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Τροπολογία 6 της Γιούτα Στάινρουκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Αντιλόπες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αν δεν κάνω λάθος, απορρίπτεται. Εντάξει. Αυτό το ελέγξουμε λοιπόν. άλλη μια υπεράριθμη ψήφος από το ΕΛΚΑ. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Τόμας Μάν. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Η νέα. Πάλι του κύριου Μάν. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Δέκα. υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 16. Υπέρ. Κατά. Άποχες Απορρίπτεται. Έλεγχο ζητείτε. Ηλεκτρονικά να ελέγξουμε παρακαλώ την τροπολογία 16. Υπέρ. Λίπερος. Α, πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. βασική D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είκοσι οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, αν δεν κάνω λάθος. «29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται». 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται». «31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την 31. Δεν ήταν και πολύ σαφές. Μάλιστα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 33 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Η 34 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Η 35 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική ε, ή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 49 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την υπαριθμό 50. Υπεράριθμη μια ψήφο από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η 51 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 52 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική H. Ήτα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 56 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Ζητείται ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 56. Θα πρέπει να επαναλάβουμε παρακαλώ την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Περισσεύει πάλι ένας από το ΕΛΚ. Απορρίφθηκε. Η 57 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η 58. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 59 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 60 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Και τώρα ψηφοφορία επί του συνόλου της ε, σχεδίου ψηφίσματος που τροποποιήθηκε υπέρ κατά Α, ηλεκτρονικά διορθώνει ο Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και πάλι ένα υπεραριθμό από το ΕΛΚ. Μάλιστα. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Προώθηση της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων. Συμβιβαστική α. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Για το σχέδιο προφορικής ερώτησης. Υπέρ. Α, μάλιστα. Ηλεκτρονικά Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του ETF. Με μυστική ψηφοφορία. Αλφαβητικά. Θα καταμετρώνται μόνο οι ψήφοι υπέρ. Είτε θα ψηφίζετε δηλαδή υπέρ, είτε δεν θα ψηφίζετε καθόλου όταν ακούτε το εκάστοτε όνομα. Πρώτος υποψήφιος Γιάν Άντερσον. Μυστική ψηφοφορία έναρξη. μόνο όσοι θέλουν να ψηφίσουν υπέρ. Αν δεν θέλετε να ψηφίσετε υπέρ, μην ψηφίσετε καθόλου. Ευχαριστώ. Πέρας. Τριάντα ψήφι υπέρ. Και πάμε στην Edith Bauer τώρα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 39 ψήφοι για την Edit Power. Jean-François Métier. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 22 οι ψήφοι για τον κύριο Μεζιέχο. Σάρα Πάρκιν. Έναρξη ψηφορία. Πέρασε. 17 ψήφοι για την κυρία Πάρκιν. Mm. Mm. Mm. Ε, Το αποτέλεσμα της ψήφου είναι ως εξής 30 ψήφοι για τον Γιάννα Άντερσον, 39 για την Bauer Edit, ε, Jean-François 22, Σάρα Πάρκιν 17. Αυτό τι σημαίνει. Ο Τάντερσον, Μπάουερ και Μεσιάχα θα είναι οι υποψήφοι μας. στη διάσκεψη των Προέδρων. Θα είναι υποψήφιοι που θα παρουσιάσουμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκαν έτσι οι ψηφοφορίες μας. Mm. Mm. Σε δύο λεπτά θα περάσουμε στην πρόταση για τους ναυτικούς. Αλλά προηγουμένως παρακαλώ θέλω ησυχία στην αίθουσα. Είναι ένα, μια πολύ σημαντική έκθεση για την Επιτροπή μας.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 Έλεγα λοιπόν ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίες των ανθρώπων που δουλεύουν σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναθεώρηση του κειμένου αυτού είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει να κάνει με πέντε οδηγίες. Έχει να κάνει με την οδηγία όσον αφορά την προστασία των ε, ναυτικών σε περίπτωση που πτωχεύσει ο εργοδότης Έχει να κάνει με την οδηγία για τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής επιτροπής ευρωπαϊκής. Υπάρχει οδηγία που φτιάχνει πλαίσιο για την ενημέρωση και την διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Έχει να κάνει με την οδηγία για την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τις συλλογικέ απολύσεις και έχει να κάνει και με την οδηγία για τα δικαιώματα των εργαζόμενων στην περίπτωση που υπάρξει μεταφορά της επιχείρησης. Πέντε οδηγίες λοιπόν έχουν να κάνουν με το κείμενο αυτό. Πρόκειται για ένα σχέδιο οδηγίας που απέτυχε στη δικιά μας ε, την ε, Επιτροπή τον Απρίλιο του 2014. Είχαμε ελάχιστο χρονικό διάστημα και ο συνάδελφος που το είχε αναλάβει, επειδή έλεγε η θητεία έπρεπε να βιαστεί πολύ. Και έτσι δεν μπόρεσε να κάνει τις διαβουλεύσεις που θα έπρεπε να είχε κάνει και οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να συμφωνήσουν. Έκτοτε, από τον Απρίλιο δηλαδή του 2014, τι έχουμε κάνει. Πρώτον, η κατάσταση τροποποιήθηκε επειδή οι κοινωνικοί εταίροι, κυρίως τα συνδικάτα και οι εφοπλιστές, οι πλειοκτήτες, δεν είχαν καταφέρει να συμφωνήσουν επί του κειμένου. Αλλά ένιωσαν ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ, ότι θα επαναρχόμασταν στην νέα θητεία. Οπότε τελικά αυτό που έκαναν ήταν διαπραγματεύσεις και κατάφεραν να πετύχουν μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των εργαζομένων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, αλλά και από την άλλη μεριά λαμβάνεται υπόψη και η ιδιαιτερότητα του κλάδου. Κάτι το οποίο χαιρέτησαν όλες οι πολιτικές ομάδες στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στις 2 Δεκεμβρίου του 2014. Εγώ πάλι θέλησα να έχω διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, συνεργάστηκα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ήδη ευθύ αρχής είχα υπόψη μου να συνεργαστώ και με τους αδέρφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες, τους κοιόδης εισηγητές, με τους οποίους είχαμε πραγματικά ιδιαίτερα επικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων. Γι' αυτό και θέλω εδώ όλους ιδιαίτερους να τους ευχαριστήσω τον Ανιέ Σιγκερχιούς, για παράδειγμα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, τον Γκερίκε από το ICR, Άλλο από τους φιλελεύθερους, από Τρίτη Γιάρικ από του Γκουε, Τζιμι Λάμπερς από τους Πράσους και την Τιάννα Πεγκίν από το EFDD. Ήταν ε, πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε όλοι τις ίδιες πληροφορίες. Ο πολιτικός μας στόχος είναι να γίνει πιο ελκυστικός ο κλάδος των ναυτικών, γιατί είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θελήσαμε να πετύχουμε το στόχο της ε, βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των συνθηκών ε, εργασίας των ναυτικών. Ευχαριστώ λοιπόν όλους ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους και τη γραμματεία βέβαια της Επιτροπής μας που μας επέτρεψαν να καταλήξουμε εδώ που έχουμε καταλήξει. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο Ζωτάλ δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να επιμείνω σε κάποιες τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί και οι οποίες περιλαμβάνουν τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Δεν την προδίδουν είναι από την τροπολογία 9. Όπου εδώ έχουμε αντιγράψει βασικά τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων χωρίς να έχουμε αλλάξει τίποτα από τη συμφωνία αυτή. Και αυτό αποτελεί πολύ σημαντική πρόοδο. Στην τροπολογία αριθμός 1 θέλουμε να υπογραμμίσουμε την οικονομική σημασία που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν τους πολλές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τροπολογία 2, ότι εδώ θέλουμε να βγούμε από καταστάσεις διάκρισης σε βάρος των εργαζομένων αυτών, των ναυτικών δηλαδή. Στην τροπολογία 3 θελήσαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι παρεκκλήσεις αυτές υπογραμμίζονται επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν χώρες που τηρούν αυτές τις παρεκκλήσεις, τις εξαιρέσεις και ότι δεν υπήρξε καμία προσφυγή. Στην τροπολογία 6 θέλουμε όλος ιδιαίτερος να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκε εργασίες των ναυτικών, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το ναυτολιακό τομέα. Η τροπολογία 7 είναι σημαντική, επειδή γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις σε περίπτωση απολύσεων, πρέπει να ενημερώνονται οι ναυτικοί, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές όταν το πλήρωμα βρίσκεται στη θάλασσα και όχι στην χώρα προέλευσης. Κυρία Πρόεδρε, λίγο πολύ αυτές είναι οι τροπολογίες που προτείνουμε προκειμένου να καταλήξουμε σε μια νέα οδηγία η οποία να μην κάνει διακρίσεις σε βάρος των ναυτικών. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Η Γιούτα Στάινμπρουκ από τους ε, σοσιαλιστές. Ναι, ο Άγνος ο οποίος ε, έχει υποχρεώσει στην εκλογική του περιφέρεια σήμερα με παρακάλεσε να μιλήσει εξ ονόματός του, ε, η κυρία Γιονγκέριους μάλλον, λέει ότι με, με το κείμενο αυτό καταφέρνουμε να προσεγγίσουμε τον στόχο μας να καταργήσουμε τις κριτικές μετα... διακρίσεις κατά των ναυτικών σε διάφορους ε, τομείς. Ε, οι κοινωνικοί εταίροι παρουσιάσανε μία συμβαστική πρόταση που θέτει τις ιδιαίτερες αξιώσεις σε ό,τι αφορά τις ναυτικές μεταφορές και όλα τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν. Η πρόταση της κυρίας Μωράν Σαρτιέρ συμπεριέλαβε αυτά που ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι για να κλείσουν τα χάσματα που υπάρχουν σήμερα και για να μπορούν να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει ίση μεταχείριση των ναυτικών. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε ως σοσιαλδημοκράτε την πρόταση αυτή. Και στο σημείο αυτό η Άκνε Γιονγκέριους θα ήθελε να ευχαριστήσει και τους κοινωνικούς εταίρους και την κυρία Σαρτιά για την εξαιρετική εργασία της. Ε, υποστηρίζουμε το στόχο της βελτίωσης των εργασιακών συνθήκων, ε, της κοινωνικής προστασίας, του καλύτερου διαλόγου μεταξύ εργαδοτών και εργαζομένων και την προώθηση της απασχόλησης στην ε, θαλάσσιες μεταφορές και ελπίζουμε με επιτυχία να στεφτεί αυτή η έκθεση που είναι προς το συμφέρον των όλων μας άλλωστε. Thank you, Ο κύριος Γκέρικε. Σας ευχαριστώ την εισηγήτρια καταρχάς, την κυρία Μωρόν Σαχτιέ, η οποία εξ αρχής έδειξε πνεύμα μεγάλης συνεργασίας. Αλλά ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο που προέκυψε μετά από στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και νομίζω ότι τελικά έχει ως αποτέλεσμα ένα ισορροπό κείμενο. Και εγώ τις τελευταίες εβδομάδες μίλησα πολύ με εκπροσώπους της βιομηχανίας, με ναυτικούς, αλλά και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις από παρακτήσεις περιοχές της Γερμανίας. Και πολλές φωνές λένε ότι η νομοθεσία για τους ναυτικούς δεν θα πρέπει να σταματάει στα εθνικά σύνορα. Η σχετική νομοθεσία χρειάζεται διασυνοριακή παγκόσμια ευρωπαϊκή προοπτική, μια άποψη που υποστηρίζει η ομάδα μου. Υποστηρίζουμε μέτρα τα οποία εξισώνουν τους ε, ναυτικούς ό,τι αφορά τις εργασιακές συνθήκες με όλους όσους εργάζονται στην ξηρά. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να δημιουργούν περί το άχθος γραφειοκρατικό ή ε, επιπλέον κόστος. Γι' αυτό λοιπόν θα ελέγξουμε και τις τραπολογίες. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι να δημιουργήσουμε κανόνες που θα, καταστούν, θα, θα καταστήσουν δύσκολο για τους ε, ναυτικούς μας να πλέουν με ευρωπαϊκές ε, σημαίες. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο στόχος μας. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί. Χρειαζόμαστε εξίσου ευέλικτους κανόνες όπως και άλλες τρίτες χώρες θα πρέπει λοιπόν να το αναγνωρίσουμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν το εργατικό δίκαιο για τους ναυτικούς να είναι εξίσου σταθερό και βέβαιο όπως και για τους υπόλοιπους και να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να παραμείνει στην πορεία της. Thank uh, from the Group. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Συμφωνώ με αυτά που είπε η εισηγήτρια για την ανάγκη και τη σημασία αυτής της οδηγίας. Γενικά, είναι καλό αυτό το σχέδιο έκθεσης. Οι κοινωνικοί εταίροι, όπως αναφέρθηκε και όλοι ξέρουμε, έχουν φτάσει σε μια συμφωνία για αυτή την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε σεβασμό για τους κοινωνικούς εταίρους και τις συμφωνίες τους, που πιστεύω ότι, και πιστεύω το κάνει η συγγήτρια, όμως σε κάποια σημεία το σχέδιο έκθεσης αποκλίνει λιγάκι από τη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων, νομίζω. Ως Κοινοβούλιο γενικά και ως Επιτροπή Απασχόλησης ειδικά, μιλάμε πολύ για τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και με αυτή την έκθεση και με αυτή την οδηγία έχουμε μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να δείξουμε απόλυτο σεβασμό για την συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Θεωρώ ότι αυτή η έκθεση είναι δοκιμή για το αν μπορούμε να σεβαστούμε πραγματικά τους κοινωνικούς εταίρους και τον κοινωνικό διάλογο ή όχι. Με βάση αυτή την γραμμή πλεύση θα κινηθώ απέναντι στην έκθεση. Βρίσκω καλό το σχέδιο έκθεσης και αδειμονώ να συνεργαστούμε περαιτέρω επί των διαφορών τροπολογιών. Ευχαριστώ. Από τους πράσινους η Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Συντάσσεται και η ομάδα μου ε, σε όλους όσους ευχαρίστησαν την εισηγήτρια. Αλλά και γενικά συμφωνούμε με αυτούς που είπαμε συμφωνούν με τις προτάσεις της ηγήτριας. Και εμείς το ίδιο. Και μάλλον μία-δυο τροπολογίες θα καταθέσουμε μόνο. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος, μια και είναι πολύ καλή δουλειά που έκανε η συγκήτρια. Η ε, Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Εμείς μόλις ξεκινήσαμε την συζήτηση από την οδηγία αυτή. Ξεκινάμε από την ιδέα ότι οι ναυτικοί πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όσους εργάζονται στην ξηρά. Δηλαδή, οι ίδιες αμοιβέ και η ίδια προστασία. Και η οδηγία αυτή πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ανάγκη να προστατεύσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας σε αυτόν τον τομέα από το κοινωνικό ντάμπινγκ. Χαιρόμαστε για τη δουλειά που έκανε η συγγύτρια σε αυτή την οδηγία. Θέλουμε με τις τροπολογίες μας να συνεισφέρουμε στις δουλειές της Επιτροπής αυτής, ούτως ώστε οι διατάξεις για τη βελτίωση της κατάστασης των ε, ναυτικών σε όλη την Ευρώπη να συνοδευτούν από την προώθηση της ε, υγείας, ε, της προστασίας, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, προστασία των ναυτικών κτλ. Νομίζω ότι μπορούμε να να κάνουμε και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε ως Κοινοβούλιο, να μην υπολοιπόμεθα από αυτό που κάνουν οι άλλοι για την προστασία των ναυτικών. Ευχαριστώ. Η προθεσμία είναι για τις ατροπολογίες 29 Ιανουαρίου, η υιοθέτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης 1η Απριλίου, ψηφοφορία στην Ολομέλεια, μάλλον Απρίλιο ή Μάιο, δοκιμαστικά το λέω. Η κυρία Λόπεθ Φοντανιέ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πράγματι. Είμαι σκιώδης συζητητής στην Αλία. Και κοιτώντα τι γίνεται στις διάφορες επιτροπές, πιστεύω ότι πηγαίνουμε στην ίδια γραμμή όλοι. Και έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει η εξαίρετη δουλειά της κυρίας Αρχιαμορτιέ, η οποία για άλλη μια φορά ετοίμασε ένα καλά ισορροπημένο κείμενο. Είναι σημαντικό και το είπαμε και χθε στην Αλία ότι η συμφωνία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς εταίρους. Με την οδηγία αυτή οι ναυτικοί θα μπορούν να αποφελούνται από τα κατάλληλα επίπεδα προστασίας που θα είναι ίδια σε όλες τις χώρες μέλη και δεν θα υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος τους σε σχέση με άλλα επαγγέλματα, κάτι το οποίο ισχύει μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταργηθούν οι εξαιρέσεις που αναφέρονται σε διάφορες νομοθεσίες και έτσι δεν θα υπάρχει και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Θέλω επίσης να επενθυμίσω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους του κλάδου. Χρειαζόμαστε νέους στον τομέα της ελίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χρήσιμο όλα αυτά. Η θέλει να πει μερικά καταληκτικά λόγια. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Εξ ονόματος της α, πολιτικής τους ομάδας. Παρα, σημείωσα τις α, παρατηρήσεις και τις ανησυχίες. Οι σκιώδεις συγητές και εγώ θα έρθουμε σε επαφή όταν χρειαστεί να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Και ενδεχομένως για να φτιάξουμε συμβιβασμούς, συμβαστικές ε, προτάσεις. Για τη Γιούτα Στάινρουκ, για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το σχέδιο οδηγίας στην ε, διαπαραταξιακή συνάντηση που κάνουμε μεταξύ συνδικάτων και κοινοβουλίου. Να περάσει το σχέδιο οδηγία και να εξεταστεί από την ομάδα εργασία αυτή ε, των συνδικάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μελών τη διοίκηση. Σα ευχαριστώ που ήσασταν τόσο επικοδομητικοί. Καταληκτικά τι να πω, ότι η συμφωνία που συνάθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που ήταν δύσκολη, δηλαδή μεταξύ πλειοκτητών και εμένων του πληρώματος, μας υποχρεώνει και εμάς τους πολιτικούς να μας πιέζει να βρούμε τα μέσα για να φτιάξουμε ένα κείμενο που θα προστατεύει τους ναυτικούς, το σύνολο των ναυτικών, στα πλοία που φέρνουν ευρωπαϊκές σημαίες. Και εγώ πιστεύω ότι είναι κρίσιμη αυτή η έκθεση, λέει η Πρόεδρος. Πάμε στο 13 της ημέρησιας διάταξης, το σημείο 13, που είναι η επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Θα δώσω το λόγο στην Αν Σάντερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους συμβούλους που με βοήθησαν και κατεύθυναν στη σύνταξη αυτής της πρώτης νομοδότησης που συντάσσω ως ε, Ευρωβουλευτής. Το κείμενο το οποίο μας ε, απασχολεί σήμερα, εξετάζουμε, το υποβάλλουμε, το εκπονούμε για την ΕΚΟΝ. Η, η ΕΚΟΝ αποφάσισε να ετοιμάσει μία έκθεση πρωτοβουλίας που θα αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Τώρα το κείμενο που μας απασχολεί σήμερα, που έχουμε μπροστά μας, το δικό μας κείμενο, αφορά το μέλλον του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Ενώ επανεκκινεί η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε όχι μόνο οικονομικό και δημοσιονομικό συντονισμό με σεβασμό των κανόνων του παιχνιδιού, όχι μόνο αυτό το μέλημα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα κοινωνικό συντονισμό για να διευκολύνουμε την κοινωνική ευημερία και να απελευθερώσουμε το δυναμικό απασχόληση στην Ευρώπη. Είμαι πεπισμένη ότι το να δώσουμε στην οικονομική διακυβέρνηση ένα πρόσωπο πιο κοινωνικό που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις, ε, την υγιή οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση, αλλά κυρίως και την απασχόληση, θα επιτρέψει στους πολίτες μας να θεωρήσουν το ευρωπαϊκό project, το project ευρωπαϊκής οικοδόμησης δικό τους. Μέσα σε αυτή την οπτική ε, σύνταξα την έκθεσή μου γύρω από δύο άξονες σε πρώτη φάση μιλάω για τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού πλαισίου και να προτείνω κάποιους τρόπους λειτουργίας του, ούτω ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό και να λαμβάνει περισσότερον υπόψη την κοινωνική διάσταση. Πρότεινα να οργανώνονται συντονιστικές συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ και του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ στα πλαίσια της υιοθέτηση των ειδικών αναχώρας συστάσεων, ούτως ώστε να προωθηθούν οι οικονομικές πολιτικές, αλλά και κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης. Επίσης, η σημασία της ένταξης κοινωνικών δικτών στον πίνακα αποτελεσμάτων του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης που προσαρτάται κάθε χρόνο στην ετήσια εξέταση της ανάπτυξης, αυτό θα σημειώσει μεγάλη πρόοδος να την υπόψη είναι η κοινωνική επίπτωση των μακροοικονομικών μέτρων. Και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ε, συνέχισης της ε, χρήσης του. Σε μια δεύτερη φάση θα ήθελα να δώσω έμφαση στις ε, ειδικέ συστάσεις που διαβιβάζονται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Πέρα από ένα πλαίσιο που τιμωρεί, σήμερα που ξεκινάει η ανάπτυξη ξανά, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα έξυπνο πλαίσιο που δίνει κίνητρα για καλές πρακτικές. Αυτή η ευκαιρία μας δίδεται μέσω της εφαρμογής συστάσεων της Κομισιόν. Είτε οικονομικές είτε κοινωνικές, θέλω να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να τις εφαρμόσουν αυτές τις συστάσεις. Δεν πρέπει να θεωρηθούν ως επιπλέον κόστος, αλλά ως επενδύσεις μακροπρόθεσμες. Φερρυπίν, καταπολεμώντας αποτελεσματικά την ανεργία των νέων μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικά και γρήγορα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων ή υποστηρίζοντας την κινητικότητα τη διασυνοριακή, ενισχύοντας Φερρυπίν το, τη δικτυακή πύλη Eures ή διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, μπορούμε πραγματικά να πάμε προς μια ανάπτυξη και απασχόληση πιο βιώσιμη στην Ευρώπη. Τώρα, πώς μπορεί να βελτιωθεί το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα βλέπω όλα αυτά. Μέσα στα πλαίσια ενός συνεχούς οικονομικού διαλόγου με όλα τα θεσμικά όργανα, εθνικά και ευρωπαϊκά, αλλά και με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τόσο ώστε να αυξηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος. Καταληκτικά, πρέπει να προλάβουμε για, και όχι να θεραπεύουμε, για να μην ξαναγνωρίσουμε καταστάσεις από τις οποίες μόλις βγαίνουμε σήμερα. Θα πρέπει να δούμε τα οικονομικά θέματα μέσα από τα κοινωνικά και την απασχόληση. Την οικονομική ανάπτυξη έτσι πρέπει να τη δούμε. Ε, θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πλήρη απασχόληση και στην κοινωνική προστασία, ούτως ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά ως όπλα ε, για μια ευημερούσα οικονομία. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά ήθελα να σας πω σήμερα το πρωί και είμαι τώρα στη διάθεσή σας για να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στη γνωμοδότηση αυτή. Όλες τις παρατηρήσεις θα τις λάβω υπόψη. Merci. Ε, Ευχαριστούμε. Το λόγο έχουν τώρα οι σκιώδει εισηγητέ, πρώτα απ' όλα από του σοσιαλιστέ, ο Σέρχιο Γουτιέρεθ Πριέτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Γι' αυτό το πρώτο σχέδιο έκθεσής της. Ευχαριστώ και για τις επεξηγήσεις που έδωσες. Ημερίζομαι πολλά από αυτά που είπε. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μια ζωτική σημασία σε έκθεση αυτή τώρα που είμαστε στην αρχή της θητείας μας. Γιατί πιστεύω ότι όντως πρέπει να αλλάξουμε το μηχανισμό οικονομικής διακυβέρνησης. Διότι είδαμε ότι από τότε που άρχισε ενισχυόμενος με το 2-pack, 6-pack κτλ. Είδαμε ότι έχουμε μια ανισορροπία ισορροπία ανάμεσα στην μακροοικονομική πολιτική και την αναγκαιότητα συντονισμού και τον, την εξέταση των επιπτώσεων που έχει. Αυτή η ισορροπία λοιπόν που υπάρχει τώρα που αξιολογούμε και αποφασίζουμε για νέες οικονομικές πολιτικές, για την ανεργία για παράδειγμα, πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Είναι αλήθεια ότι θα είχα προτιμήσει η έκθεση αυτή να μην είναι μόνο μία άποψη, διεκδικούμε κάτι. Εμείς η Επιτροπή Απασχόλησης εδώ και καιρό διεκδικούμε. Και πρέπει να βάλουμε στο ίδιο επίπεδο τα κοινωνικά και την απασχόληση, στο ίδιο επίπεδο με τα οικονομικά. η άποψη της Επιτροπής μας θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με εκείνη της Οικονομικής Επιτροπής, για παράδειγμα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μηχανισμός συντονισμού που άρχισε πριν από λίγα χρόνια είχε έναν βασικό στόχο και αυτός ήταν να συνδέσει τις πολιτικές των ευρωπαϊκών θεσμικών ε, οργάνων με την εφαρμογή τους στις χώρες ώστε να πετύχουμε τους στόχους το 2020. Είμαστε πολύ μακριά από αυτούς όμως γιατί ακριβώς ο μηχανισμός συντονισμού δεν λειτουργήσε για να πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν οι μηχανισμοί. Κάτι μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, να υπάρχουν κοινέ συνεδριάσεις κοφίν και έψκο. Αν όμως στη συνθήκη δεν μπορούμε να βάλουμε αυτά που θέλουμε, αν δεν μπορούμε τις οδηγίες και τα λοιπά να τα βάλουμε στο ίδιο επίπεδο, αυτές που αφορούν δηλαδή την απασχόληση και αυτές που αφορούν την οικονομία, ε, δεν θα πετύχουμε. Οι κοινωνικοί δείκτες, όταν αξιολογούμε τα οικονομικά μέτρα τα οποία εγκρίνονται εδώ και στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να είναι ισχυροί, να είναι επαρκείς και να έχουν κάποιες συνέπειες. Γιατί τι είδαμε από τότε που εγκρίθηκε η δέσμη των εξοδιών. Όταν ένα κράτο μέλος απομακρύνεται από το έλλειμμα ή από το χρέος, υπάρχουν συνέπειες. Αν όμως ένα κράτος μέλος έχει 25% ενεργεία, έχει δείκτες φτώχειας πάνω από 20%, έχει κοινωνικά δράματα, δεν γίνεται τίποτα. Και εκεί θα έπρεπε να υπάρχουν συνέπειες. Και εκεί υπάρχει οικονομική ανισορροπία και κυρίως μεγάλα προσωπικά δράματα πρέπει να υπάρχει κάποια πολιτική συνέπεια, πρέπει να υπάρχει κάποια αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει κάποιο έλεγχο και παρακολούθηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν γίνεται όμω. Πρέπει επίση να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα. Εδώ με το μηχανισμό διακυβέρνησης δεν τον βοηθάμε αν δεν βάλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή όταν σχεδιάζονται οι πολιτικές που αφορούν τους πολίτες. Ειλικρινά «Ναι, το πιστεύω αυτό. Και με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Εντάξει, θέλουμε διοργανική συμφωνία, εννοείται μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, ακριβώς για να είμαστε στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο. Γιατί είναι σαφές ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί με μη δεσμευτική γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι που παγώνει την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μεγαλύτερη νομιμότητα δηλαδή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο Κοινοβούλιο το οποίο πρέπει να συμμετέχει στην οικονομική διακυβέρνηση και το σχεδιασμό τη. Τέλο τα εθνικά κοινοβούλια. Κοιτάξτε, έχουμε πετύχει με το μηχανισμό συντονισμού οι υπερπολογισμοί των χωρών μελών να στέλνονται πρώτα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πριν να έχουν εγκρεθεί οριστικά από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όμως, τι γίνεται με την Εθνική Κυριαρχία. Δεν περνούν ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να κόψετε εκεί ή αλλού στην εκπαίδευση, στην απασό, δεν ξέρω πού, ή στις συντάξεις. Μα δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς και τα Εθνικά Κοινοβούλια είμαστε που εκπροσωπούμε την Ευρωπαϊκή Κυριαρχία, την κυριαρχία των πολιτών. Εμείς πρέπει να έχουμε άποψη για αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα. Τέλος είναι πολύ σημαντικό στους μηχανισμούς αυτούς αναθεώρησης της διακυβέρνησης να υπάρχει χώρος και για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Νιώθουν αποκλεισμένοι. Και όταν οι εκπρόσωποι των πολιτών και οι πολίτες αυτοί καθ' αυτοί νιώθουν αποκλεισμένοι από έναν μηχανισμό, τότε μπορούμε να περιμένουμε άνοδο του λαϊκισμού και των ακραίων τάσεων. Κάποιοι προσπαθούν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια να φτιάξουν κάποιες ομάδες όπου να συμμετέχουν οι πολίτες. Μα χρειάζεται επίσημο διάλογος, ανοιχτός, σοβαρός, που να επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να δουλέψουμε. Είναι καλό σημείο κίνηση η έκθεσή σα. Συμφωνώ με τα πρώτα που άκουσα από την εισηγήτρια και κατά τη γνώμη μου μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε κάτι πολύ βασικό μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Κωνσταντέψκη από το ECR, παρακαλώ. Σκιώδης εισηγητής του ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για, την, ε, για το σχέδιο έκθεση. Πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία περιλαμβάνονται στο πρώτο σχέδιο της έκθεσης, ιδιαίτερα στο δεύτερο τμήμα τη έκθεση και συμφωνούμε με τα στοιχεία αυτά τα οποία με βρίσκουν και προσωπικά πολύ σύμφωνο, απλά αμφιβάλλω ε, για το πρώτο τμήμα της ε, έκθεσης, για παράδειγμα στο σημείο 1 συμπαριλάβατε μια θετική αξιολόγηση της διαδικασίας συντονισμού μέχρι σήμερα, συντονισμό των ε, οικονομικών πολιτικών δηλαδή ως τώρα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί ένα θέμα για το μακρινό μέλλον, για το απότερο μέλλον συμφωνούμε όλοι. Αλλά η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ω τώρα νομίζω ότι μάλλον αρνητική θα έπρεπε να είναι και αυτό θα έπρεπε να αποτυπώνεται στην έκθεσή σα. Επίση, στην ομάδα μα δεν πιστεύουμε όλοι ότι αυτόματα υπάρχει συσχετισμός, σύνδεση μεταξύ του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, κρίσιμη σημασία θα έλεγα, να τονίσουμε το τι ακριβώς εννοείται στο σημείο 2 του σχεδίου σας, ε, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η υποβατικότητα όλου, όλης της εργαλειοθήκης, όλων των μέσων που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τούδε. Θα ήθελα να αναφερθώ και στον προηγούμενο ομιλητή και αυτό που αναφέρεται στο σημείο 10 της έκθεσής σας. έχουμε την πρόθεση να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Είναι θέμα δημοκρατικής νομιμότητας ή δημοκρατικού ελλείμματος, όπως το δει κανείς. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει μόνο να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό θα μεταφραστεί σε αποδυνάμωση των εθνικών κοινοβουλίων και του ρόλου τους. Ε, μας απασχολούν τα κοινωνικά δικαιώματα εδώ στην Επιτροπή μας και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στα εθνικά κοινοβούλια υπάρχει κόσμος που γνωρίζει σε βάθος τι, γνωρίζει, τι χρειάζεται ακριβώς ο κόσμος στην εκλογική τους περιφέρεια και από δημοσιονομικής απόψης και άλλα ζητήματα. Αν όλα αυτά μεταφερθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό το μόνο που θα πετύχει είναι να αυξήσει την αίσθηση δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη. Συμφωνώ εκεί που αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει σε θέματα συντονισμού της οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν πιστεύω ωστόσο ότι η συμμετοχή μας εδώ θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να κλείσει το δημοκρατικό έλλειμμα, το δημοκρατικό χάσμα. Δεν θα πρέπει να μιλάμε λοιπόν για εμβάθυνση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να καταστήσουμε το εργαλείο αυτό πιο αποτελεσματικό αλλά περιορισμένο. Ευχαριστώ κύριε Γκασνοτεύσκη και τώρα να δώσω το λόγο στο σκιώδη των ε, φιλελευθέρων, την κυρία Όλα Τόρνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή γνωμοδότηση. Καλύπτει πολύ σημαντικά σημεία για την οικονομική διακυβέρνηση και το πλαίσιο αυτής. Και συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια που υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας ε, για το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και μιλάει για τη συνέχιση της ε, διαβούλευσης. Συμφωνώ ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για τις ειδικές συστάσεις αναχώρα και τη βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, συμφωνώ με την άποψη της συζητήτης για πιο στενό οικονομικό διάλογο μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν και επομένως αύξηση της, οικονομικής, της δημοκρατικής λογοδοσίας. Θεωρώ ότι ο ρόλος μας ως η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι να βρούμε και να συνεχίσουμε μια έτσι προσπάθεια να συμπεριλάβουμε και την διάσταση της απασχόλησης. Η Επιτροπή μας έχει μια ατζέντα που είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη ατζέντα οποιασδήποτε άλλη επιτροπή. Τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιε θέσεις, όπως είπε και η συγκήτρια, θα πρέπει να συνεχίσουμε την οικονομική εξυγίανση. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην οικονομία, γιατί αυτό είναι θεμέλιο για την ιδιωτική επεν... Ε, τις ιδιωτικές επενδύσεις και είναι η θεμελιώδης, η ακροκονιές λίθος για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτό αντανακλάται στην γνωμοδότηση και με ικανοποιεί. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένη με το σχέδιο έκθεση. Μπορεί να στείλω λίγε τροποποίησεις που θα τονίζουν τη σημασία τη ε, συνέχιση τη προσπάθεια τη οικονομική εξυγίαση για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και τον σημαντικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ακριβώ για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσει στην Ευρώπη. Εργασία στην Ευρώπη. Από την Κουένα Σούπερ αλλά δεν είναι εδώ. Αλλά πάμε στην, τότε στην κυρία Βάνα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την εισηγητρία για τις ε, ερμηνείες που έδωσε. Αλλά θα πρέπει να πω ότι εμείς ως πράσινοι δεν συμφωνούμε με την κατεύθυνση και με τις παρατηρήσεις που γίνονται εδώ στην έκθεση. Και επειδή η ανάλυση, το είπαν άλλωστε και οι προηγούμενοι ομιλητέ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ε, αν ξεκινάμε από την πρώτη παράγραφο που μιλάει για την ευφυή ανάπτυξη που προκαλείται, νομίζω ότι τα αριθμητικά στοιχεία μας διαψεύδουν ικτρά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την εντύπωση αυτή. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά άλλα σημεία, τη διατύπωση. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις επιτροπές μας. Μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιοτικέ ε, θέσεις εργασίας. Εδώ μιλάμε μόνο για ανάπτυξη και μόνο για θέσεις εργασίας το έγγραφο αυτό. Άρα θεωρώ ότι ιδιαίτερα η δική μας επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει ότι μιλάμε για παραπάνω πράγματα και όχι μόνο για τα μυστικότητα. Μιλάμε και για του στόχου τη Ευρώπη 2020, για την κλιματική αλλαγή, την καταπολέμηση τη ένδυα, την ισότητα. Όλοι αυτοί είναι στόχοι για του οποίου οι επενδύσεις και οι διαφορετικέ ε, αλλαγές, οι οποίε συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να λάβουν υπόψη όμω και τι ε, πτυχέ αυτέ. Οι κοινωνικέ επενδύσει, οι επενδύσει σε δημόσιε υπηρεσίε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσει. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν μπορεί να ε, έχει αυτό ο στόχο περαιτέρω απορρίθμιση, αλλά την ε, καταπολέμηση της φτώχειας, του περιθωριοποίησης, την... Ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα ενισχύσουμε στο κείμενο, όπως και την παράγραφο για τους κοινωνικούς δείκτες. Θέλω να την τονίσουμε. Θεωρώ ότι είναι θέμα κλειδί. Τονίζω ότι με... μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι αναφέρονται τα μοντέλα βέλτιστων πρακτικών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά θεωρώ ότι και η περιφερειακή εταίροι θα πρέπει να αναφερθούν γιατί εκεί αναπτύσσονται και θα πρέπει να ανταλλαχθούν τα συστήματα βελτιστών πρακτικών. Αυτό που μας ε, λείπει, το είπαν άλλωστε και κάποιοι προηγούμενοι συνάδελφοι, είναι η δημοκρατική λογοδοσία και η συμπερίληψη στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, η κοινωνία των πολιτών δηλαδή, μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Χθε το συζητήσαμε αυτό επισταμένο σε ό,τι αφορά και την ετήσια έκθεση ανάπτυξη. Η προηγούμενη επιτροπή είχε θέσει ω στόχο την μεγαλύτερη συμπερίληψη τη κοινωνία των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σε ό,τι αφορά τι κατευθυντήριε γραμμέ. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να το ζητήσουμε στην έκθεση. Και μέχρι τι 30 Ιανουαρίου λοιπόν θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίε στο πνεύμα αυτό που σα ανέφερα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Η Λαούρα από το EFTD. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη συνάδελφο για την ανάλυση της. Το κίνημα των πέντε αστέρων έχει να κάνει κάποιες επικρίσεις και κάποιες διευκρινήσεις πάνω στο κείμενο αυτό. Καταρχάς, γιατί το να έχουμε αυταρέσκεια το να μιλάμε τόσο θετικά για το ρόλο της οικονομικής διακυβέρνησης νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο, δεν λαμβάνει υπόψη ότι πολύ συχνά η οικονομική διακυβέρνηση στις χώρες γίνεται μια επιταγή, μια πίεση ε, ασφικτική μάλιστα και δεν επιτρέπει μια συμμετοχή και την ανάπτυξη και αντί να προλάβει τις ανισορροπίες, κυρίως τις ε, κοινωνικές, τις ενθαρρύνει και τις πολλαπλασιάζει. Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση για εξορρόπηση του, του προϋπολογισμού, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά, εντάξει, αλλά θα έπρεπε να εμπλακούν και οι κοινωνικοί εταίροι σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ξεχνάμε λιγάκι τη διάσταση των πολιτών και την πραγματική ζωή που διάγουν. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για την ανεργία των νέων. Σύμφωνοι. Αλλά να, αντιμετωπίσουμε και τις άλλες μορφές ανεργίας. Δεν έχουμε μόνο την ανεργία των νέων, έτσι. Μάλιστα είναι πιο ανησυχητική και πιο πιεστική η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τη μακροχρόνια ανεργία, κυρίως που οφείλεται και που ε, λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών. Το να αντιμετωπίσουμε τώρα την ανεργία των νέων. Για να την αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να μιλήσουμε κυρίως για τη δημιουργία εργασίας, θέσεων απασχόλησης. Μ' αρέσει να μιλάω για την ενίσχυση επίσης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συχνά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν χρηματοδοτεί, δεν δίνει πίστοση στις ΜΜΕ, αλλά μόνο τα μεγάλα προγράμματα και τα μεγάλα project. Και αυτό που φτάνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ψυχία. Τώρα, για τη διασυνοριακή κινητικότητα. Λέμε ότι είναι ευκαιρία ας μετακινηθούμε, ας φύγουμε. Υπάρχουν δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Ωραιότατα. Να στείλουμε τους νέους να δουλέψουν σε άλλη χώρα. Αλλά πότε εμείς θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Θα αδειάσουμε λέει, τις χώρες που έχουν κρίση, θα τις κάνουμε ερήμους. Γιατί υπάρχουν θέσεις απασχόλησης σε άλλες χώρες. Εγώ θέλω να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα μας, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να δώσουμε ευκαιρίες. Γιατί η κινητικότητα καλή είναι, αλλά η κάθε χώρα νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει στο εσωτερικό της θέσεις απασχόλησης. Γιατί αλλιώς θα έχουμε ένα τμήμα της Ευρώπης έρημο, ακατοίκητο, γιατί θα υπάρχουν θέσεις. Και όλοι θα πάνε αλλού. Κάποιος είπε ότι πρέπει να προλάβουμε και όχι να θεραπεύουμε. Δυστυχώς, η αρρώστια μας είναι σοβαρότατη. Θα μ' άρεσε η πρόληψη. Αλλά τώρα πρέπει να θεραπεύσουμε κιόλας λιγάκι. Γιατί ζω σε μια χώρα άρρωστη, στη ρίζα της άρρωστη. Θα μιλήσουμε για πρόληψη όταν θεραπεύσουμε την αρρώστια που μας τρώει τώρα. Την αρρώστια των χωρών όταν θα έχουμε δώσει φαΐ στο τελευταίο ε, πεινασμένο παιδί που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Όταν θα έχουμε, ε, διορθώσει την καταστροφική κατάσταση των, του κράτους πρόνοια σε διάφορες χώρες. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για την θεραπεία των προβλημάτων των φτωχών χωρών. Ε, ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Σάντερ έχει το λόγο και πάλι να δώσετε κάποιες απαντήσεις ή τι σκέφτεστε για αυτά που ακούσατε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρεμβάσεις σας, τις πολύ θετικές. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων για διάφορα σημεία. Είτε πρόκειται για την ε, δημοκρατική νομιμότητα, είτε για το διάλογο, είτε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, αν πρέπει να ενισχυθεί ή όχι, με ποιο τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε. Όλα αυτά είναι θέματα για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί. Ήδη τώρα για να ολοκληρώσω θέλω να μιλήσω για την ημερήσια διάταξη. Στην Επιτροπή Οικονομικών Θέσεων μεταφέρθηκε το θέμα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας για να ανταλλάξουμε απόψεις εδώ. Οπότε τώρα κοιτάζω με την γραμματεία της δικιάς μας Επιτροπής να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε τις τροπολογίες ενώ αρχικά δεν προβλεπόταν αυτό. Θα ήταν καλό, ενδιαφέρον να το κάνουμε για όλους μας. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 30η Ιανουαρίου και εννοείται ότι είμαι στη διάθεσή σας ολονών για να ανταλλάξουμε ακόμα και διμερώς αν θέλετε απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ και τίποτα άλλο. Είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η προθεσμία είναι η 30 Ιανουαρίου και θα εγκριθεί στις 26 Φεβρουαρίου η έκθεσή σας εδώ στην Επιτροπή μας. Αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές εννοείται ότι θα σας ανακοινωθούν. Τρεις και τέταρτο θα αρχίσουμε με το κεφάλαιο 2 της συνεδρίασης αυτής το δεύτερο τμήμα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Τρεις και τέταρτο και πάλι.